την ομάδα μάλλον των Δημοκρατών, των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών έχω λάβει ε, ορισμούς σε επιτροπές και αντιπροσωπείες που δημοσιεύονται στα συνοπτικά πρακτικά. Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση θεωρούνται ως εγκεκριμένες αυτές οι προτάσεις. Η Επιτροπή Ιστορικής